Αγαπητοί συνάδελφοι, επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Παρακαλώ να καθίσετε. Έχουμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ε, της εκλογής των αντιπρόεδρων του Κοινοβουλίου. Ο αριθμός των ψηφισάντων είναι 702. Λευκάη Άκυρα 41 661 ψήφισαν απόλυτη πλειοψηφία 331 Οι υποψήφοι πήραν τους ακόλουθους ψήφους, τις ακόλουθες ψήφους. Κυρία Μαγκίνος, 618, εκλέγεται. Πέντρο Σίλβα Περέιρα, 556. Εκλέγεται. Ονορεύολε Βίλαντ. Ο κύριος Βίλαντ, 516 εκλέγεται. Μπάρλεϊ 516 εκλέγεται. Ονορεύολε Κάρας. Ο κύριος Κάρας 477 εκλέγεται. Ονορεύολε κύριος Κόπατς. 461 εκλέγεται, κυρία Κόπατς. Ονορεύολε Κλάρα Ντόμπρευ, 402 ψήφοι, εκλέγεται. Χαραντσόβα, με 395 ψήφους εκλέγεται. Συνάδελφος Μπέρ, 363 ψήφους εκλέγεται. Γιάροκα, 349 ψήφια εκλέγεται. Η κυρία Χαουτάλα, 336 ψήφια εκλέγεται. Αυτή είναι η υποψήφοι που πέτυχαν την απόλυτη πλειοψηφία. Ο κύριος Παπαδημούλης, 303 ψήφους. Κολάγια, 237 ψήφους. Κρασνοντεύσκη 169. Καστάλτο 143. Ουτασάρη 135 ψήφους. Μπιτσότο 130 ψήφους. Οι συνάδελφοι αυτοί δεν εξελέγησαν. Φυσικά θα ήθελα να συγχαρώ τους συναδέλφους για την εκλογή τους. Αλλά για το Προεδρείο του Κοινοβουλίου έχουμε ακόμα τρεις έδρες και επομένως πρέπει να προχωρήσουμε σε νέα ψηφοφορία. Θα περάσουμε σε μια δεύτερη ψηφοφορία. Λοιπόν, αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, θεωρούν ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι υποψηφιότητες της πρώτης ψηφοφορίας. Υπάρχουν παρατηρήσεις? Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, οι υποψηφιότητες της ε, πρώτης ε, ψηφοφορίας τηρούνται. Η δεύτερη ψηφοφορία θα γίνει στις μισή, προκειμένου να σφραγιστούν τα ψηφοδέλτια και θα τα ξαναπούμε εδώ στην αίθουσα για την ψηφοφορία. Ραντεβού λοιπόν στις ε, μισή, Διακόπτη τη συνεδρίαση. sì, lo, eh, se mi chiedi la parola lo dici e così... Eh, però qui non abbiamo i nomi. Allora, colleghe e colleghi, la seduta... Συνάδελφοι, επαναλαμβάνει εταιρεία συνεδρίαση πρέπει να γίνει η δεύτερη ψηφοφορία για την εκλογή τριών επιπλέον αντιπροέδρων. Ο κύριος Τζάνι έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να διαβιβάσω ότι η ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία αποφάσισε να αποκλείσει μία από τις δύο υποψηφιότητες ε, της ε, κυρίας ε, Χουταζάρη θα παραμείνει μόνο υποψηφιότητα της κυρίας Μπιτζότο. Ωραία, το σημειώνουμε και επομένως τώρα πρέπει να ξανατυπώσουμε τα ψηφοδέλτια και για να γίνει αυτό θα συνεχίσουμε με την ψηφοφορία στις 7. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.